από πλευράς ε, των αστυνομικών αρχών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε, κύριε Χέντεγκάρτ. Έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος ε, ε, και ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Για τις, με τις ψηφοφορίες για τους ΛΟΑΔΑ στην Αφρική. Έχουμε ένα κοινό σχέδιο ψηφίσματος πέντε πολιτικών ομάδων και ψηφίζουμε πρώτα την παράγραφο 3. Ψήφι ΠΕΡ. Α, συγγνώμη, είναι κατά τμήματα, σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι ΠΕΡ. Δεύτερο, κατά, συγγνώμη, εποχές εγκρίνεται. Δεύτερον, ΠΕΡ Κατά, αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο. Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία για την παράγραφο 2, το δεύτερο τμήμα. Τώρα αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα ψήφου υπέρ. Κατά και αυτό θέλει έλεγχο, μάλλον η ίδια πλειοψηφία θα είναι, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Παράγραφος 16, στο αρχικό κείμενο, Ψήφιπε. Κατά. Και αυτό θέλει επαλήθευση. Μπορεί να φαίνεται η ίδια πλειοψηφία αρχής ψηφοφορία τώρα, αλλά είναι μικρή διαφορά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. Απορρίπτεται με διαφορετική πλειοψηφία παρόλα αυτά. 18 ψηφί υπέρ. Κατά. Και αυτό θέλει έλεγχο. η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία, ή αν και μεγαλύτερη, απορρίπτεται. Η παράγραφος 20. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. Η τελική σκέψη όμικρον λατινικό, το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Ε, πρώτον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ονομαστική είναι η τελική ψηφοφορία, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι από πέρας. Εγκρίνεται 33-24. Ερχόμαστε τώρα στο ψήφισμα για την ελευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία. Έχουμε και εδώ ένα κοινό ψήφισμα. Πέντε πολιτικών ομάδων. Και υπογράφει και ο κύριος Πάσκα. Ψήφι υπέρ του συνόλου κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στα ψηφίσματα για την αναγκαστική άμβλωση στην Κίνα. Έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος έξι πολιτικών ομάδων που υπογράφει ο κύριος Πάσκα. Η τροπολογία 3 στην παράγραφο 2 Ψηφίπε κατά έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και καταπέφτει το αρχικό κείμενο. Αν κατάλαβα καλά. Μετά την παράγραφο 7, δύο τροπολογίες, η ψήφη υπέρ, τις δύο, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη Δέλτα, η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ερχόμαστε τώρα στο σύνολο του ψηφίσματος, όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Η κυρία Βεζιά θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δαπανούμε υπερβολικό χρόνο για την προετοιμασία των κατεπηγόντων σε συνεδριάσεις που αποσκοπούν στην εξέβρεση συνένεσης μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Ε, το θεωρώ λοιπόν λυπηρό να υπάρχουν κάποιες συγκυριακές ε, πλειοψηφίες από διάφορες ομάδες που καταθέτουν ε, τροπολογίες που ούτε στα κοινά ψηφίσματα ούτε ε, στη συνεργασία σε αυτές τις κοινές συναντήσεις που είχαμε κάνει είχαν αναδυθεί καταργώντας τελικά τους συμβιβασμούς οποίους προσπαθούμε να καταλήξουμε δραματικό και είναι και καταστροφικό για την κοινή δουλειά που συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στο ημικύκλιο. Ιδίω για την τρίτη μάλλον εννοεί πέμπτη απόγευμα, που δεν είμαστε και τόσο πολλοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βερζιά. Υποθέτω ότι και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε που είναι τόσο προσιλωμένε και αφοσιωμένε συμφωνούν. Τα πρακτικά θα διανεμηθούν προ έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση και αν